οπαδούς ε, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επιτρόπο Κάλλας και κλείνοντας ε, να αναφέρουμε ότι έχουμε έξι ε, ψηφίσματα και θα κάνουμε κατευθείαν την ψηφοφορία. Περνάμε στο πρώτο θέμα της ψηφοφορίας. Επτά ψηφίσματα για τις συγκρούσεις στα σύνορα Ταϊλάνδης και Δεν έχουμε προτάσεις για τα κοινά ψηφίσματα και θα ήθελα να ψηφίσουμε συνολικά υπέρ. Κατά. Άποχες. Το ψήφισμα λοιπόν ομόφωνα εγκρίθηκε και περνάμε τώρα στο ψήφισμα για την ιεμένη θα ποινή εναντίον ανηλίκων ατόμων, ιδιαίτερα η περίπτωση του Μοχάμετ Ταχέρ Θαμπέτ Σαμούμ. Έξι ψηφίσματα, ένα κοινό ψήφισμα έχει διαμορφωθεί. Έχουμε κάποιες τροπολογίες. Καταρχάς, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται η τροπολογία και περνάμε στην τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Άποχες. Επίσης εγκρίνεται και περνάμε τώρα στην τροπολογία σε τμήματα για την παράγραφο 1. Ποιος είναι υπέρ του αρχικού κειμένου. Κατά. Άποχες. Μία αποχή λοιπόν έτσι αποφασίζεται και περνάμε τώρα στο κείμενο. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Για την ιδεολογική σκέψη α για το 1 υπέρ κατά άποχες και αυτό εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη συνολική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά άποχες το ψήφισμα λοιπόν και αυτό εγκρίνεται και περνάμε στο τελευταίο ψήφισμα για την Ουγγάντα, δολοφονία του Ντέβιτ Κάτο και εδώ έχει προκύψει λοιπόν πλέον κοινό ψήφισμα. Θα ψηφίσουμε καταρχά την παράγραφο 6 σε δύο τμήματα. Καταρχάς το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Πάμε σε χωριστή ψηφοφορία στην παράγραφο 8 του αρχικού κειμένου. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Άποχες. Και αυτό εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την παράγραφο 12 του αρχικού κειμένου. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψήφισετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Και περνάμε τώρα στη συνολική ψηφοφορία για το τροποποιημένο κείμενο με νομική ονομαστική συγγνώμη, ε, ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορία. Αν ψήφισατε όλοι, πέρας ψηφοφορία. Ομόφωνα και με μία ψήφο αποχής εγκρίνεται το ψήφισμα. Και έχω κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω από πλευράς Συμβουλίου έλαβα και την θέση του Συμβουλίου και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τρεις μήνες προθεσμίες από την αυριανή ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου έχει τη διάθεση του το Κοινοβούλιο